Okay. Please, uh, let's start our work because we are late. ξεκινήσουμε επειδή έχουμε αργήσει. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα εξ ονόματος της Προέδρου να κάνω ορισμένες ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η ψηφοφορία που είχε προβλεφθεί για αύριο αναβάλλεται για τις 7 Ιουνίου. Δεύτερο, ο τριμερής διάλογος, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, για εθνικούς και περιφερειακούς λογαριασμούς, ε, που έλαβε χώρα στις 16 Μαΐου και ο δεύτερος τριμερής διάλογος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 1η Ιουνίου. CRD4, trialogue is going on. Διάλογος βρίσκεται σε εξέλιξη, τίποτε άλλο, τίποτε άλλο. Trialogue took place on 20... 2, τελευταίο τριμερής διάλογο στι 24 Μαου. Αυτά είχα να σα πω από πλευρά ανακοινώσεων. Α περάσουμε τώρα στην πρώτη έκθεση σχέδιο γνωμοδότησης, εξέταση των τροπολογιών. Αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης έχει σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας καταναλωτικής πίστης και ήθελα να σας πω τα αποτελέσματα από τη μελέτη των τροπολογιών. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συνέταξαν αυτές τις τροπολογίες και, τις και την συνάδελφό μας από τη γραμματεία, την κυρία Τζένιφερ Λάγκ, που με βοήθησε για να εξετάσουμε τις τροπολογίες και να καταλήξουμε σε ορισμένους συμβιβασμού. Προτείνω τρεις, τρεις συμβαστικές τροπολογίες και πρώτα απ' όλα έχω την ε, συμφωνία των συναδέλφων. Η πρώτη συμβαστική τροπολογία αφορά το δικαίωμα που των πελατών να ενημερώνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, δηλαδή της ε, ε, καταναλωτικής πίστης προσυμβατικές και στη διάρκεια της σύμβασης να ενημερωθούν σχετικά με τους κινδύνους που αναλαμβάνουν τη στιγμή που συνάπτουν μια σύμβαση καταναλωτικής πίστης σε ξένο, σε συνάλλαγμα και θα πρέπει συνεπώς να ενημερώνονται και οι πληροφορίες να είναι εξατομικευμένες, κατανοητές κτλ. Εδώ καλύπτουμε την τροπολογία 1 του κ. Μόλτσερ, την τροπολογία 2 και 12 του κ. Ντιμπέκερ, την τροπολογία 3 του κ. Γίγκορντ, 4 της ε, κυρίας Μακάρθη. Η δεύτερη συμβαστική τροπολογία αφορά την ιδέα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αξιολογήσουν τον κίνδυνο που συνιστά ο δανεισμός σε συνάλλαγμα. Επίσης, να αξιολογήσουν την ικανότητα του καταναλωτή Ε, να αντιμετωπίσει τις δοκιμάνσεις ε, στις τιμές εναλλάγματος και την αποπληρωμή του δανείου φυσικά. Αυτή η συμβατιστική τροπολογία καλύπτει επίσης πολλές τροπολογίες που έκαναν ο κύριος Μπέκερ 13, 14, Δίγκολντ, 15 κυρία Σουίνμπουρν, ο κύριος Ντεμπέκερ 10, 11 και πάλι ο κύριος Δίγκολντ 29 και 31. κατατέθηκαν διάφορες τροπολογίες ή μάλλον ξέρετε τι προτείνω στο σχέδιο γνωμοδότησής μου προτείνω δύο πράγματα που απερίφθησαν όμως αυτές οι δύο προτάσεις από διάφορους συναδέλφους και εντάξει το καταλαβαίνω έχουν δίκιο η πρώτη πρότασή μου λοιπόν ήταν ότι δεν πρέπει να δεχόμαστε μια, ένα, μια καταναλωτική πίστη που υπερβαίνει την πενταετία όσον αφορά περίοδο αποπληρωμής και ο κύριος και ο κύριο Ντιμπέκερ ε, προτείναν να διαγραφεί αλλά εγώ πιστεύω ότι η κυρία Σφρίμπορν έκανε μια καλή πρόταση. Γι' αυτό και υποστηρίζω την πρόταση της κυρίας Σφρίμπορν. which um, που καλεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να λάβουν υπόψη τους σοβαρά τις περιπτώσεις χωρίς δανείων με διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε ετών στο πλαίσιο των καταναλωτικών δανείων προκειμένου να διασφαλίζεται ότι εξυπηρετούν το βέλτιστο συμφέρον του εν λόγω καταναλωτή. Αυτή η πρόταση με βρίσκει σύμφωνο και κατά συνέπεια προτείνω να καταψηφιστεί η πρόταση Μόλτσον και Μπέκτα αλλά να δεχθούμε την τροπολογία που προτείνει η κυρία Σουίνμπουρν. Το ίδιο αφορά και την πρότασή μου ε, να μην συμφωνήσουμε όταν υπάρχει μια οικογένεια ενός ατόμου μόνον και γίνεται στεγαστικό δάνειο, της χορηγείται στεγαστικό δάνειο, πάλι υπάρχουν διάφορες ε, τροπολογίες που προτείνουν να διαγραφούν, αλλά η κυρία Σουίμπουρν μας έκανε μια καλή πρόταση, μια καλή τροπολογία και γι' αυτό συμφωνώ με αυτή την τροπολογία της, η οποία είναι... financial Ή τα χρηματιστικά ιδρύματα να δώσουν κατανοητική πίστη μόνον όταν υπάρχουν εγγύσεις, κατάλληλες εγγύσεις για να εξασφαλιστεί ένα ικανό επίπεδο κινδύνων και για τους δύο, για τα δύο μέρη. Επίσης υπάρχει μια ε, συμβιβαστική ε, τροπολογία C που καλύπτει την τροπολογία 25 του κ. Γκίφουντ και 26 του κυρίου Νικολάου Χουντή. Αυτή η συμβαστική τροπολογία αφορά το δικαίωμα του πελάτη, του καταναλωτή δηλαδή, να ενημερώνεται σχετικά με το κόστος των συμπληρωματικών υπηρεσιών, καθώς και για το δικαίωμα του καταναλωτή να επιλέγει βοηθητικές υπηρεσίες που παρέχονται από εναλλακτικού προμηθευτές ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όχι εκείνα που χορηγούν το δάνειο, να γίνεται διάκριση μεταξύ βοηθητικών υπηρεσιών που είναι ουσιαστικές ε, για τον πάροχο του δανείου και τέτοιου είδους βοηθητικές υπηρεσίες οι οποίες είναι προαιρετικές για τον δανειζόμενο. Port, ε, amendments, ε, του κυρίου Μπέικορ, υπαριθμών 5, 8, 28 και με βρίσκουν σύμφωνο αυτές οι τροπολογίες, καθώς και του κύριου Κάρινς 27, Μακάρθη 30 και Γκίγκολντ 6, υπαριθμών 6. Η τροπολογία υπαριθμών 6 και 32. And again, miss, uh, Πάλι, κυρία Σουίμπορν, τροπολογία 18 ε, και 23. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες που προτείνει ο κ. Νικόλαος Χουντής. Uh, uh, δεν συμφωνώ με ορισμένες από αυτές τις τροπολογίες. Η μία που προτείνει ο κ. Χουντής καλύπτεται από μια συμβαστική τροπολογία. Αλλά δεν συμφωνώ με όλες. Θα τα δούμε στην ψηφοφορία βεβαίως. Επειδή αυτές οι τροπολογίες είναι όπως οι συμβουλές που δίνονται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δεν νομίζω να είναι ο σωστός χώρος εδώ να αναφέρονται αυτά τα θέματα. Είναι γενικότερα θέματα που αφορούν αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είχα να σας πω. Αν η κυρία Μερκάρτη είναι εδώ ή κάποιος που την εκπροσωπεί, σκιώδη συγγήτρια, παρακαλώ. Εδώ ήταν η κυρία Μακάρθη, αλλά έφυγε για λίγο. Πάντως γενικά στηρίζει τις ε, συμβιβαστικές σας προτάσεις και πιστεύω λοιπόν ότι καταλήγουμε σε ένα αποτέλεσμα πολύ ενδιαφέρον και ισορροπημένο. Αυτά είχα να πω εξ ονοματός της. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ για τη συνεργασία στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Μας βρίσκουν σύμφωνος και δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε να καταλήξουμε επί αυτών ε, οι διάφορες ομάδες. Ένα ή δύο θέματα θέλω να αναφέρω μόνο. Το ένα αφορά τη διαφήμιση και τις ε, πρακτικές marketing. Είναι ρυθμιζόμενες ε, οι αγορές σε μεγάλο βαθμό, αλλά υπάρχουν κάποιες πρακτικές που προσελκύουν ε, τους καταναλωτές. είδα μια διαφήμιση με email που έλεγε ότι αν σας απέρριψε, αν ε, στην τράπεζα. Μην ανησυχείτε, θα, και θα, σας, θα έρθετε σε εμά και θα σας δώσουμε οπωσδήποτε καταναλωτικό δάνειο. Ε, δεν θέλω να απαγορευτούν τελείως αυτές οι πρακτικές βέβαια και αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε μέσα από τη γνωμοδότηση το πρόβλημα, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή να πιέσει την Κομισιόν να ε, λύσει το θέμα αυτό της παραπλανητικής ψευδούς διαφήμισης. Επίσης, στη 18 και 23 της κυρίας Σουίνμπορν, Ιδιαίτερα στην 23 αναφέρονται οι εγγυήσει και καμιά φορά είναι δύσκολο ε, ε, να το λύσουμε αυτό στην καταναλωτική πίστη. Στην ενυπόθηκη εκεί το, η εγγύηση είναι το σπίτι. Στην καταναλωτική πίστη όμως τι θα κάνουμε. Θα δώσουμε τη τηλεόραση, τη συσκευή της τηλεόρασης ως εγγύηση. Δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Οπότε διστάζω λίγο να δώσω την υποστήριξή μου στις δυο αυτές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κι εγώ να επαναλάβω τους επένους των άλλων συναδέλφων. Ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία. Θα στηρίξουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες σας και ευχαριστούμε για τη στήριξη δύο ακόμη τροπολογιών. Νομίζω ότι ε, συμβάλλουμε σωστά για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στην οδηγία καταναλωτικής πίστης και νομίζω ότι τώρα πρέπει να κάνουμε λόμπι στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, ούτως ώστε να τα συμπεριλάβει όλα αυτά. Και σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα επιτύχουμε και την υποστήριξη της Επιτροπής ΙΜΚΟ εδώ. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίσης, όπως αναφέρατε, συμπεριλάβατε μία από τις τροπολογίες μου στην τρίτη συμβιβαστική πρόταση, επομένως την ενισχύω. Ε, είναι σωστό αυτό που είπατε καταρχήν. Δηλαδή ο λόγος που δεν ε, εγκρίνεται, δεν υιοθετείτε τις άλλες τροπολογίες, αλλά θα σας έλεγα θα άξιζε τον κόπο ενδεχομένως να, τους, να τις ξαναδείτε. Δεν είναι συμβουλές που δίνουν οι οικονομικοί όμιλοι. Είναι νομίζω ένα πρόβλημα που πιάνει την ουσία του θέματος και την οποία έχετε αντιληφθεί ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ε, δεν αναφέρομαι στις γενικές κατευθύνσεις, στις γενικές σκέψεις που περιέχουν κάποιες τροπολογίες γιατί πράγματι μέσα από τη γνωμοδότηση δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα το πώς οι τράπεζες δίνουν τα καταναλωτικά δάνεια αλλά ε, και ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η καταναλωτική πίστη είναι πώς βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο και θα ήθελα να σας πω κύριε Πρόεδρε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ τραγική σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω της αδυναμίας να αποπληρωθούν τα καταναλωτικά δάνεια στις τράπεζες. Το ιδιωτικό χρέος στη χώρα μου αλλά όχι μόνο στη χώρα μου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αντιλαμβάνομαι ότι η γνωμοδότηση δεν μπορεί να το λύσει. Παρά τα αυτά από αυτές τις τροπολογίες που δεν ε, υιοθετείται θα, σας, θα επαναλάμβανα μόνο με τίτλους ότι η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου φορέα που θα έδινε συμβουλές στους πολίτες σχετικά με τη διαδικασία αυτή θα ήταν βοηθητική. Ξανασκεφτείτε το, δεν είναι κάτι το φοβερό δηλαδή που ανατρέπει λογικές και ούτω καθεξής. Επίσης το θέμα για την πρόορη, εξόφληση των δανείων χωρίς να επισύρει αυτό ποινές. Και το τρίτο και τελευταίο για να μην σας κουράσω είναι αυτό που είπα και στην αρχή υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με τα καταναλωτικά δάνεια που δεν μπορούν να αποπληρωθούν λόγω ύφεση και περικοπών και θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί προτάσεις που και οι τράπεζες να μην έχαναν σε ρευστότητα και ταυτόχρονα να προσαρμόζονταν οι δόσεις του δανείου στις περιορισμένες αποδοχές που έχουν αρκετοί εργαζόμενοι σε αρκετές χώρες. Αυτά κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την προσοχή που δείξατε στις τροπολογίες που κατέθεσα.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 θα περιοριστώ σε ένα σχόλιο, αφού ευχαριστήσω πάλι όλους τους συναδέλφους για τις τροπολογίες τους. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Νικόλα Οχουντή. Καταλαβαίνω πολύ καλά που αναφέρεστε και στη Ρουμανία παρόμοια είναι η κατάσταση. Όταν πρότεινα να σταματήσει ο δανεισμός σε οικογένειες με καταναλωτική πίστη, όταν ζητούσαν εγγύηση τα σπίτια τους και τώρα πολλές πετάχτηκαν έξω από το σπίτι τους οικογένειες από τις τράπεζες γιατί δεν μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειο, βέβαια ενοχλήθηκα πολύ και κατάλαβα ότι δεν μπορώ να στηρίξω μια τέτοια ε, πρόταση να σταματήσει ο δανεισμός ε, σε τρα... Ε, από τράπεζες σε οικογένειες ε, όταν ε, το σπίτι είναι το μόνο ακίνητο που διαθέτουν και το μόνο περιουσιακό του στοιχείο. Στις 7 Ιουνίου θα γίνει η ψηφοφορία. Στην Επιτροπή 18 Σεπτεμβρίου, εολομέλεια ε, τον Οκτώβριο, στις 7 Ιουνίου θα συζητήσουμε περαιτέρω. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σχέδιο γνωμοδότησης με συντάκτη τον κύριο Φιλίπ Λάμπερτς για πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές. Κύριε Λάμπερτς, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γνωμοδότηση, δεν θέλω να χάσουμε πολύ χρόνο, παρόλο που το θέμα είναι σημαντικό, μια και μιλάμε για αυτά τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας κυρίως, που μπορούν και θα έπρεπε να παίξουν κέριο ρόλο στην ε, οικονομική ανάπτυξη. Μιλάμε πολύ για την μεγέθυνση και την ανάπτυξη. Είναι ένας τομέας λοιπόν εδώ που μπορεί να δημιουργήσει αξία ε, με βιώσιμο τρόπο αν χρησιμοποιήσουμε το μέσον καλά. Μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπής, είναι η ήτρε αρμόδια επί της ουσίας και αυτό μου επιτρέπει να σχολιάσω ότι κάποιες τροπολογίες των συναδέλφων δεν ε, ανήκουν στην Επιτροπή ΕΚΟΝ αλλά στην Επιτροπή ΙΤΡΕ. Γι' αυτό δεν τη συμπεριέλαβα σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον, αφού δεν ενδιαφέρουν το έργο της Επιτροπής μας, είναι πολύ τεχνικές και πολύ λεπτομέρειες. Έχοντας ε, δει τις τροπολογίες που λάβαμε για τα άρθρα και τα προσαρτήματα και τα... τις αιτιολογικές σκέψεις, είναι ομόφωνες με την έννοια ότι όλες είναι χρήσιμες ε, ως προσθήκες στο κείμενο και θα πρέπει να είμαστε ευτυχείς διότι δεν είναι αντιφατικές. Τώρα, τα βασικά σημεία εδώ είναι η σύνδεση μεταξύ της δημιουργίας αυτών των ενεργειακών υποδομών και των χωρών σε κρίση στο πρόγραμμα. Θέλουμε να υπάρχει μια σύνδεση εδώ για να αποδείξουμε ότι πράγματι τα δίκτυα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των χωρών σε κρίση και εδώ εισάγουμε την ιδέα αυτή ε, της ταχείας διαδικασίας ανάπτυξης αυτών των έργων σε, ε, σε αυτές τις χώρες. Δεύτερον, αυτό που θέλουμε είναι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για, την, για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την ιεράρχηση των έργων να είναι πιο διαφανείς από ό,τι είδαμε μέχρι τώρα. Και γι' αυτό μεταξύ άλλων μιλάμε για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις στα κριτήρια. Φοβάμαι ότι κάποιοι από εσάς δεν στηρίζουν τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και θέλω να το καταλάβω αυτό γιατί λέτε ότι βαραίνει πολύ η πρόταση. Όμως αυτός είναι ένας τρόπος ώστε το Κοινοβούλιο να ε, δει ποια είναι τα κριτήρια και μια και μιλάμε για ιεράρχηση στις δαπάνες δημοσίου χρήματος νομίζω ότι χρειάζονται σαφή κριτήρια που θα ελέγχονται από το Κοινοβούλιο. Δεν είναι κακό αυτό. Ίσως πιστεύουν μερικοί ότι η κατεξουσιοδότηση πράξη είναι πολύ βαριά διαδικασία, αλλά αν έχετε εναλλακτική, βεβαίως θα την ε, θεωρήσω ευπρόσδεκτη. Κάτι άλλο είναι να υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτών και της υπερκείμενης ευρωπαϊκής στρατηγικής που είναι η EU 2020. Περισσότεροι από εμά συμφωνούμε ότι θέλουμε μεγαλύτερη συνέπεια στην χρήση των ενωσιακών πόρων και το σημείο αναφορά είναι η στρατηγική 2020, Ευρώπη 2020 και θέλουμε να υπάρχει συνέπεια μεταξύ αυτών των διευρωπαϊκών δικτύων και των προτεραιοτήτων του 2020. Το ίδιο για τα διαρθρωτικά ταμεία. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Μία ιδέα που έχουμε εισαγάγει εδώ και που θα θέλαμε να εφαρμόζεται ευρύτερα στον προϋπολογισμό της Ένωσης είναι μια ρήτρα που προβλέπει αναθεώρηση όταν το κόστος του έργου ξεπερνά το αρχικά υπολογισθέν κατά 20%. Το ποσοστό μπορούμε να το συζητήσουμε. Αν όμως έχουμε ε, μεγάλη υπέρβαση κόστους, τότε θα πρέπει να επανεξετάσουμε το έργο για να βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε εδώ ε, μια ανεξέλεγκτη κατάσταση που απορροφά συνεχώς κονδύλια. Τι άλλο για να δούμε. Νομίζω ότι ένα άλλο θέμα που δεν συγκέντρωσε η ομοφωνία είναι η ψήφος ε, με πλειοψηφία και όχι ομοφωνία. Συνήθως ομοφωνία ισχύει, αλλά βέβαια ε, μπορεί εν προκειμένου να μην είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος ε, λήψης αποφάσεων. Σταματώ εδώ για να ακούσω τους Σκιώδης, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω για την συμβολή τους. Ο κύριος Λάγκεν που είναι και Σκιώδης. Συγγνώμη. Μόλις ήρθα και δεν άκουσα όλα αυτά που είπε ο συνάδελφος, με συγχωρείτε. Είναι ε, πολλή ώρα πρέπει να περιμένουμε για τα σανσέρα από το 15ο. Μιλήσαμε για τις συμβαστικές τροπολογίες και πρέπει να πω ότι συνολικά η ομάδα ΕΛΚ μπορεί να συμφωνήσει με τα περισσότερα σημεία. Ζητήσαμε σε ένα σημείο τμηματική ψηφοφορία και το γενικότερο ερώτημα είναι αν ε, οι προδιαγραφές που έχουν τύχει επεξεργασία εδώ στις συμβιβαστικές τροπολογίες, εάν θα δώσουν περαιτέρω εξουσίες στην Κομισιόν. Στη συμβιβαστική Α ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε εκεί. Επίσης, ποια θέματα θα ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο, αλλά νομίζω, μην έχοντας ακούσει βέβαια τον συνάδελφο, μπορώ να πω ότι ε, μπορούμε να έχουμε σε μεγάλο βαθμό ε, ενιαίο κατάλογο ψηφοφοριών. Στη συμβιβαστική α υπάρχουν δύο σημεία στα οποία ζητούμε, στο 3α και στο 4α ζητούμε τμηματική ψηφοφορία. Ε, θα το δούμε και στις λεπτομέρειες. Ε, σκεφτόμαστε να ψηφίσουμε υπέρ και η συμβιβαστική Β είναι εντάξει. Η δυσκολία εν μέρη ήταν ότι τώρα που ήταν η πεντηκοστή δεν μπορέσαμε να δουλέψουμε και ο κατάλογος ψηφοφοριών μόλις τώρα παρελήφθη οπότε δεν μπορούσαν να γίνουν προηγουμένως διαπραγματεύσεις. Συνολικά όμως η ομάδα ΕΛΚ μετά από ε, ε, εκτενή έλεγχο και διαβουλεύσεις θα μπορέσει να συμφωνήσει στη μεγάλη πλειοψηφία των θεμάτων. Ευχαριστώ. Η κυρία Περέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ε, κυρία Άννη Ποδηματά, σιώδη συγγήτρια, βρίσκεται σε μια άλλη Επιτροπή και μου ζήτησε να διαβάσω την ε, θέση της ε, ως ε, σκιώδης συγκήτρια. Να ευχαριστήσω τον κύριο Λάμπερτ αλλά και τους σκιώδης συνεισηγητές. Πιστεύουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό και με σημαντική προστεμένη εργασία για την Ήτρε που είναι και η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Καλωσορίζουμε τις νέκατες γραμμές σχετικά με τις ενεργικές υποδομές, κάτι το οποίο συμβάλλει στα βασικούς στόχους της ενεργικής πολιτικής, διασφαλίζει την βιωσιμότητα, την αραγωνιστικότητα κλπ. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη αυτών των υποδομών αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλή, χαμηλής έντασης διοξιδίου του άνθρακου. Ε, Ζητάμε να υπάρξουν κανόνες για τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος. Το σχέδιο γνωμοδότησης του κ. Λάμπερτ και οι συμβαστικές τροπολογίες που προτείνονται βελτιώνουν το αρχικό κείμενο και θα στηριχθεί από την πολιτική μας ομάδα. ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να αποδοθεί τροπολογίες που αφορούν τους περιβαλλοντικούς στόχου και τους ενεργειακού στόχου τη Ευρωπαϊκή ένωση, όπως επίσης και τη συμβολή της Ένωσης στη στρατηγική για ανάπτυξη και απασχόληση. Ακούσαμε την παρουσίαση του εισηγητή και θα θέλαμε να πούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι χώρε που αντιμετωπίζουν δυσκολίε. Θέλαμε να τονίσουμε πολλέ σημαντικέ προσθήκε που έλειπαν από το αρχικό κείμενο, όπω η αποφυγή οδήποτε στρέβλωση του ανταγωνισμού, ειδικά ανάμεσα σε σχέδια τα οποία στοχεύουν στις αυτές προτεραιότητες. Δεύτερον, την υπέρβαση των δυσκολιών για, κατά την χρηματοδότηση και την διασφάλιση ότι η υλοποίηση των ε, ενεργειακών υποδομών για την επίτευξη των στόχων χρειάζεται να λάβουμε υπόψη και την σύνδεση των ε, νησιωτικών ε, περιοχών με την σύνδεσή τους με υπόλοιπε χώρε ε, σε ό,τι αφορά τη σύνδεση με το, για, την, για το ηλεκτρικό ρεύμα. Για μια ακόμα φορά ευχαριστώ την εισηγητή, τον εισηγητή και τους συνεισηγητές για τη σύμβολή τους. Αυτό που σας διάβασα είναι η στάση της κυρίας Ποδηματά. Ευχαριστώ κύριε Φερέρα. τους Κυλακάκης. Θα μιλήσω εξ του κ. Σκυλακάκη που δεν μπορεί να παραστεί σήμερα. Ε, συμφωνούμε με τον παρατήρηση σχετικά με τα πράξεις κατεξοδότηση. Η ομάδα μας όμως ε, θεωρεί ότι μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να ε, παρεμποδιστεί. Αυτή είναι η μοναδική το μοναδικό σχόλιο του κ. Σκυλακάκη και θα σταματήσω σε αυτή την παρέμβασή μου εδώ. Ο κ. Τόμας Χέντελ, σκιώδης, δεν παρευρίσκεται. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να το λόγο. Κύριε Λάγκεν. Πότε θα μας δώσει ο εισηγητής ε, τον οριστικό κατάλογο ψηφοφοριών, κύριε Λάμπερτς. Αν ψηφίσουμε αύριο, θέλουμε να ξέρουμε τις λεπτομέρειες από τώρα. Ναι, υπάρχει αυτή η ερώτηση. Έτοιμοι είμαστε, περιμένουμε τη γραμματεία να, ε, να τον αποστείλει τον κατάλογο. Έτοιμος είναι. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο και να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο. Πρόκειται για μία έκθεση. Η κυρία Ρόβη Κράτσα είναι η συγκίτρια. Hmm? Who is θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό εάν και εφόσον έρθει η συγκίτρια. Τώρα τι κάνουμε. Ο κ. Κλίντς είναι παρόν. Εντάξει. Η κυρία Πίτη Κάινεν ε, απουσιάζει. Και αυτή. Okay. We have to take a break, unfortunately, for... Να διακόψουμε για 10 λεπτά, δυστυχώς. 10 λεπτά διάλειμμα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 Okay, meeting starting again. Next... Επαναλαμβάνεται η συνεδρίασή μα Επόμενη έκθεση είναι η έκθεση σχετικά με την ελκυστικότητα των επενδύσεων στην Ευρώπη. Η συγγήτρια, η κυρία Ρόδη Κρατσά. Παρακαλώ, για το λόγο. <laughs> Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι δεύτερη φορά που συζητούμε για την ε, έκθεση αυτή. Την πρώτη φορά είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω τους στόχους και το περιεχόμενο της έκθεσης και να ανταλλάξουμε απόψεις με τους συναδέλφους. Τώρα ερχόμαστε σε, με βάση πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Ε, είχα περίπου περισσότερο ίσως από 100 τροπολογίες. Ε, προσπάθησα με την καλή συνεργασία των ε, σκιωδών ε, εισηγητών που τους ευχαριστώ θερμά και για την πολύτιμη συμβολή τους αλλά και για την καλή τους διάθεση να φτάσουμε σε ένα συνεκτικό κείμενο άρα να κάνουμε καλές συμβιβαστικές τροπολογίες. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα νέα στοιχεία που οι συνάδελφοι έφεραν με τις τροπολογίες τους, όπως ε, η βάση, η ανάγκη για μια καλή βιομηχανική, συγκροτημένη βιομηχανική πολιτική στην Ένωση που έχει υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια. Ε, άλλα θέματα που σήγαγαν οι συνάδελφοι είναι το θέμα, των, το, η σημασία του τομέα για επενδύσεις της πράσινης ανάπτυξης ε, ο σεβασμός των ε, κοινωνικών περιβαλλοντολογικών κριτηρίων ε, στην, προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με εμπορικούς εταίρους ανά τον κόσμο. Θέμα πολύ σημαντικό διότι εξασφαλίζει τις συνθήκες για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν μπορούμε να αποφύγουμε το κοινωνικό, το περιβαλλοντολογικό ντάμπινγκ σε διεθνές επίπεδο ε, ε, άλλα θέματα είναι το θέμα η σημασία της παιδείας ε, οι επενδύσεις στην παιδεία, γενικά οι επενδύσεις, ο τομέας των δημοσίων επενδύσεων, η σημασία του, ιδιαίτερα η παιδεία αναφέρθηκε από συναδέλφους και έχει ενταχθεί στις, συμβαστικές τροπολογίες. πιστεύω ότι έχουμε καταλήξει σε ένα κείμενο συνεκτικό, ε, χωρίς ε, ιδιαίτερες επαναλήψεις, απόλυτα δεν μπορούμε να το αποφύγουμε ποτέ. Και επίσης ήθελα να ευχαριστήσω και τους συντάκτες γνωμοδοτήσεων στην Επιτροπή Ήτρε και στην Επιτροπή Ρέτζι για τις ενδιαφέρουσες απόψεις τους στην κατάσταση ψηφοφορίας που σας έχει υποβληθεί ε, σε πολλές παραγράφους έχω αρνητικό πρόσημο ακριβώς διότι ε, είναι ενδιαφέρουσες ιδέες αλλά περιλαμβάνονται ήδη στο αρχικό κείμενο της έκθεσής μου ή στις τροπολογίες των μελών της ομάδας μας που έχουν ήδη ενταχθεί μέσα στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Ε, ε, αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Πιστεύω ότι στέλνουμε ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει μια πολιτική για τις επενδύσεις τις ξένες και τις εγχώριες και να μην είναι μια οριζόντια διάσταση αφημένη στις πολιτικές χωρίς να αποτελεί ένα στόχο στρατηγικής. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Ε, και πιστεύω ότι όλες οι διαστάσεις των πλεονεκτημάτων που έχουμε και πρέπει να αναδείξουμε των αδυναμιών που πρέπει να αντιμετωπίσουμε νομίζω ότι βγαίνει σε αυτό το, το πλαίσιο που δημιουργήθηκε με, μαζί με τις συμβαστικές τροπολογίες και σε μεμονωμένες τροπολογίες που έχω πρόσημο αρνητικό στην πρότασή μου είναι ε, διότι περιλαμβάνονται ή επικαλύπτονται από άλλες έννοιες που ήδη έχουν ε, προταθεί. Αυτό είναι τις γενικές γραμμές η προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Um, I'm Ευχαριστώ. Οι σκιώδεις έχουν το λόγο. Η κυρία Κλέβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να καλωσορίσω την ε, έκθεση της συγγήτριας αναφορικά με και την ενθυστικότητα των επενδύων στην Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί σε κάθε συνεδρίαση. Θεωρώ ότι μέσω των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί έχουμε πετύχει τον αρχικό στόχο και έχουμε ενισχύσει περαιτέρω το κείμενο και θα αναζητήσουμε συμβαστικέ λύσεις. Να πω ότι οι περισσότερες τροπολογίες μου τώρα αποτελούν τμήμα των συμβαστικών τροπολογιών και ευχαριστώ τον κυρία Κράτσα και του συνεργάτε της τα τελευταία χρόνια ε, στο Κοινοβούλιο, ειδικά στην ε, ομάδα των σοσιαλιστών, ζητούσαμε μια νέα στρατηγική για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την δημιουργία καλύτερων ε, ποιοτικά θέσεων για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε από την κρίση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση θα αποτελέσει ένα έναυσμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον της πολιτικής επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο επιθυμεί φυσικά και η κυρία Σιγητή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βόρφ Κλίντς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια για την εκ νέου παρουσίαση της έκθεσης με την οριστική μορφή. Δεν ήμουν στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων, ε, είχα εκπροσωπηθεί από άλλο συνάδελφο, αλλά ε, και ε, με εκπροσώπηση Σάρων Μπόλς και είπε τότε και για λογαριασμό μου ότι είμαι θετικά διακείμενος στο μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης. Τρεις τροπολογίες κατέθεσα μόνο που τις θεωρούσα σωστές γιατί αφενός ήθελα να βεβαιωθώ και να φροντίσω ότι αν συγκρίνουμε την Ευρώπη με τις ΗΠΑ, στη ρύθμιση ε, των αγορών πρέπει να έχουμε ίσους κανόνες ανταγωνισμού. Επίσης η πρόσβαση στις αγορές θα είναι εφικτή και θα διευκολύνεται και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε επενδύσεις να ε, διευκολύνονται και για αυτές τις μικρές ε, εταιρείε και επιχειρήσεις. Και επίσης τρίτον ήθελα να πω ότι η ελκυστικότητα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρου επένδυσης επηρεάζεται και από την ε, δυσμενή δημογραφική μας εξέλιξη και ότι και εδώ πρέπει να κάνουμε κάτι για να ενισχύσουμε την ελκυστικότητα της Ευρώπης. Από τις 100 περίπου κατατεθήσεις τροπολογίες, ήδη η συγγήτρια το είπε, πολλές είναι αδιαμφισβήτητες, θεωρώ, και χωρίς πρόβλημα θα καλυφθούν από συμβιβαστικές τροπολογίες Ορισμένες θεωρώ ότι πάνε υπερβολικά μακριά, διότι όχι τόσο επί της ουσίας έχω πρόβλημα, αλλά επειδή θεωρώ ότι δεν είναι ο χώρος αυτής της έκθεσης ο κατάλληλος για να αναφερθούν τα προβλήματα αυτά, όπως η προηγούμενη συνάδελφος που μίλησε για επενδύσεις από το δημόσιο τομέα, δημόσιες επενδύσεις. Χρειάζεται λίγη προσοχή εδώ, γιατί το public spending οι κρατικές δαπάνες ή οι δημόσιες δαπάνες ήταν πάρα πολλές το τελευταίο διάστημα, οπότε είμαι λίγο επιφυλακτικός. Γενικά όμως μπορώ να συμφωνήσω με τις συμβιβαστικές τροπολογίες και είμαι βέβαιος ότι αύριο η έκθεση κατά την ψηφοφορία θα συγκεντρώσει μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκίγκολτ είναι ο επόμενος κοιόδης. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για αυτή την έκθεση. Καταθέσαμε ορισμένε τροπολογίες. Βασικά, αυτό που επιθυμούμε είναι να υπογραμμίσουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη, και αυτό περιλαμβάνει και την ανάπτυξη των ε, ξένων άμεσων επενδύσεων, δεν είναι αυτός σκοπός. Αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε αυτό το τομέα για να υπάρχει η σωστή μορφή οικονομικής ανάπτυξης για να είναι πιο πράσινες οι βιομηχανίες μας και να περιοριστεί η κατανάλωση ε, των μη ανανεώσιμων πηγών ε, ενεργείας. Γι' αυτό ε, χρειαζόμαστε πολλές επενδύσεις και μια ισχυρή πολιτική για να υπάρχουν και πολλές ξένες επενδύσεις και να αυξηθούν οι επενδύσεις στην οικονομία γενικά. Πράγμα το οποίο συμβαδίζει απόλυτα με την ατζέντα της πράσινης οικονομικής ανάπτυξης. Η μελέτη δείχνει πολύ καλά τι μας κατευθύνει ε, για να υπάρχουν ε, ισχυρές επενδύσεις. Και μάλιστα, και γι' αυτό το λόγο θα έλεγα, προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε περισσότερο αυτή την έκθεση, προτείνοντας ε, να υπάρχουν πολλά δημόσια αγαθά σε τομείς όπως τις υποδομές, αλλά και την παιδεία και ε, την κοινωνία, επειδή η κοινωνική ειρήνη είναι πολύ σημαντική για να έχουμε ένα θετικό επενδυτικό κλίμα. Μετά, η μακροοικονομική σταθερότητα είναι ουσιαστική σημασία για να εξασφαλιστούν σωστέ συνθήκε για επενδύσει και η, το γεγονός ότι υπάρχει αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη οδηγεί σε μείωση των επενδύσεων. Επίσης πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια επιθετική πολιτική, επενδυτική πολιτική στον τομέα ε, τη της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, της των πόρων και της αντικατάστασης ε, του ε, φυσικού αερίου και του πετρελαίου από ΑΠΕ. Και πιστεύουμε επίσης ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα πρέπει να μην βλέπει κοντόφθαλμα ε, τα θέματα, ε, το οποίο δεν ευνοεί απαραίτητο τις επενδύσεις, αλλά να υιοθετήσει μια μακρόπνοη προοπτική. Γι' αυτό το λόγο ο χρηματοπιστωτικός κλάδος θα πρέπει να επαναρρυθμιστεί. Επίσης πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί επειδή αν τα κράτη-μέλη ανταγωνίζονται για επενδύσεις, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην καταστρέψουν την παροχή δημοσίων αγαθών από τον οποίο θεμελιώνονται επενδύσεις. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι ο ανταγωνισμός για τις επενδύσεις μπορεί να έχει και θετικές πτυχές. Παράλληλα όμως θα πρέπει να είναι ένας τίμιος αγώνας, ένα τίμιο παιχνίδι, ε, όταν έχουμε να κάνουμε με ε, κίνδυνο ανταγωνισμών κυρίως όσον αφορά την φορολόγηση των κινητών συντελεστών παραγωγής, αλλά και κυρίως όσον αφορά του ε, τα, τους, κανόνες του περιβάλλοντος και κοινωνικού κοινωνικούς κανόνες. Γι' αυτό ορισμένε τροπολογίες και συμβατικές τροπολογίες τελικά, αλλά δεν έχουμε ακόμα δει το, την λίστα της ψηφοφορία. Γι' αυτό δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια θα είναι η ε, τελική μορφή της έκθεσης και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι γνώμες των άλλων επιτροπών. Ίσως έγινε κάποιο λάθος με τον κατάλογο της ψηφορίας, δεν ξέρω, αλλά καλό θα ήταν να δούμε τον κατάλογο, τη λίστα και εν πάση περιπτώσει χρειάζεται να δούμε τον κατάλογο με τις τροπολογίες και την ψηφοφορία για να τοποθετηθούμε τελικά, για να αποφασίσουμε πώς θα ψηφίσουμε τη συνολική έκθεση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να πω δύο λόγια. Ε, παρά το γεγονός δεν είμαι σκιώδης εισηγητής για αυτό το θέμα, θα ήθελα να πω δύο λόγια παρόλα αυτά για τις επενδύσεις στην Ευρώπη και την ελκυστικότητα των επενδύσεων στην Ευρώπη. Η ελκυστικότητα των επενδύσεων στην Ευρώπη έχει σχέση με την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. Υπάρχουν ορισμένα εμπόδια που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ίδια. Κυρίως το υψηλό επίπεδο φορολόγησης είναι εμπόδιο στις επενδύσεις. Επίσης, ε, η χαμηλή αποδοτικότητα των επενδύσεων στην Ευρωζώνη κυρίως. Θα τρομάξει, θα αποθαρρύνει ορισμένου επενδυτέ αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα. Θα ήθελα επίση να υπενθυμίσω και την σημασία που έχει η ανταγωνιστικότητα. Κάθε φορά που μιλάω για ανταγωνιστικότητα, ο κόσμο πιστεύει ότι μιλάω για μια αφηρημένη, έννοια που δεν έχει και κανένα νόημα. Αλλά η ανταγωνιστικότητα, κύριε Πρόεδρε, είναι το γόνιμο έδαφος για να φτιάξει κανείς ένα περιβόλι. Και σε αυτό το περιβόλι χρειάζεται κανείς γόνιμο ε, έδαφος, χώμα καλό αν θέλουμε να αναπτυχθούμε. Λοιπόν, η αμεταγωνιστικότητα είναι αυτό το γόνιμο έδαφος. Αλλά δεν έχουμε γόνιμο έδαφος και ξεραίνεται ο κήπος μας και μαραίνονται τα λουλούδια μας επειδή η ανταγωνιστικότητά μας υπονομεύεται. Και εμείς συμβάλλουμε σε αυτό. Για παράδειγμα, ε, εισάγοντας αυτό το, το, φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Λέμε τώρα ότι θέλουμε ξένο κεφάλαιο. Αλλά τα ξένα κεφάλαια φεύγουν από την Ευρωζώνη μαζικά. Εγκαταλείπουν τα κεφάλαια και θέλουμε να τα επαναφέρουμε στην Ευρωζώνη. Και τι κάνουμε, επιβάλλουμε έναν φόρο χρηματοπιστωτικών, ε, συναλλαγών. Λοιπόν, δεν θα επανέλθουν τα κεφάλαια έτσι όπως είπε ο κ. Κλίνστ, ε, ε, τι πρέπει να κάνει την Ευρώπη, συμφωνώ ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε πολλούς τομείς. Το άλλο, η πλάνη που δημιουργούμε εμείς λέγοντας ότι χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις στο δημόσιο τομέα, ε, σε έργα υποδομών και ούτω καθεξής. Δεν είναι κακό αυτό φυσικά. Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται στην Ισπανία. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν έχει κατασκευάσει τόσα όσο η Ευρώπη. Κατά κεφαλή είναι η Ισπανία, είναι η χώρα που έχει τους περισσότερους, ε, τους περισσότερους αυτοκινητοδρόμους και έχει ανεργία 25% και μεταξύ των νέων ανεργία 50%. Λοιπόν, δεν πρέπει να δημιουργήσουμε την αυταπάτη ότι ξοδεύοντας περισσότερα έργα υποδομής τότε θα λύσουμε και όλα τα προβλήματα. Γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα όταν μιλάμε για ελκυστικότητα επενδύσεων στην Ευρώπη και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλικοί προς επενδύσεις και κυρίως να υπάρχει ανταγωνισμός στους φόρους και όχι, ε, ανταγωνισμός, όχι εναρμόνιση στους φόρους, διότι ο ανταγωνισμός στη φορολόγηση είναι που μειώνει τις επενδύσεις και αποτρέπει τους επενδυτές. Ευχαριστώ. <laughs> Uh, Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ανοίγει ε, η συζήτηση. Ζητεί κάποιο το λόγο. Όχι, από ό,τι βλέπω. Οπότε δίδω πάλι για μια τελευταία λέξη στο λόγο στην κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους και συζητητέ εισηγητές που σήμερα παρόντες ε, ανέπτυξαν τις απόψεις τους. Είναι αλήθεια ότι έπρεπε να βρούμε και εγώ μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης των επενδύσεων, των δημοσίων επενδύσεων, ε, του, impact που έχουν επενδύσει ε, στο περιβάλλον, στην ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης που ήταν οι ευαισθησίες από κάποιες πολιτικές ομάδες και το φιλικό περιβάλλον των ιδιωτικών επενδύσεων που ήταν ευαισθησία άλλων ομάδων. Πιστεύω ότι καταφέραμε μια ισορροπία στην έκθεση. Θέλω να πω καταρχάς για τον κύριο Γκίγκολτ ότι η λίστα ψηφοφορίας έχει έλθει από χθε το μεσημέρι. Και επειδή δεν είχαμε αντίδραση από την πολιτική σας ομάδα, την ξαναστήλαμε σήμερα το μεσημέρι. Μπορείτε να το τσεκάρετε με τους συνεργάτες σας, κύριε συνάδελφε. Ε, και ε, βασικά πιστεύω ότι η έκθεση αναδεικνύει τη σημασία που έχει να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας γιατί ένα έδαφος, ένα έδαφος ε, έφορο για επενδύσεις και επενδύσεις εννοούμε και ξένες και εγχώριες κύριε Επί, και ξένες και εγχώριες επενδύσεις όχι μόνο ξένες διότι έχουμε ανάγκη να ενθαρρύνουμε και την επενδυτικότητα των Ευρωπαίων επενδυτών να μην βρίσκουν ενδιαφέρον να πηγαίνουν σε άλλες περιοχές του κόσμου από την Ευρώπη. Λοιπόν, πιστεύω ότι αναδεικνύονται με τη συμβολή των συναδέλφων αυτές οι προκλήσεις και παρουσιάζεται ένα ισορροπημένο, μια ισορροπημένη πρόταση και πάλι σας ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία της συζήτησης που μας δώσατε. Ευχαριστώ. Η ψηφοφορία αύριο. Αύριο θα γίνει η ψηφοφορία. Αύριο. Και τώρα προχωρούμε στο σχέδιο γνωμοδότησης που ακολουθεί. Έχουμε δύο εισηγητές, τον κύριο Βολφ Κλίνς και την κυρία Πιτικάινεν. Είναι τροπολογίες για δύο διαφορετικές οδηγίες. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις, γιατί καταρχήν θα αναφερθώ και στις δύο εκθέσεις πριν ε, αναφερθώ σε αυτές μία-μία. Πολύ σημαντικό θέμα και στις δύο εκθέσεις είναι σε ποιο βαθμό οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν από εμάς τις ε, εργασίες τους να τις κοινοποιούν στη χώρα, αναχώρα δραστηριοποίησης. Επίσης, πέραν τούτου, σε ποιο βαθμό οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να δίνουν υποχρεωτικά πληροφορίες για τα επιμέρους έργα τα οποία ε, υλοποιούν στις χώρες. Στις δικές μου προτάσεις, καταρχήν, ε, σκέφτηκα μια λύση πακέτο, γιατί βλέπω να υπάρχει μια σχέση μεταξύ της υποχρεωτικής συμπερίληψης διαφόρων επιχειρήσεων, δηλαδή την εξορυκτική βιομηχανία ε, που ε, κάνει εξόριξη πετρελαίου ή αερίου ή άλλων πρώτων υλών και αν δούμε τον αριθμό, αν διευρύνουμε τον αριθμό των επιχειρήσεων για να συμπεριλάβουμε σε μια ακραία περίπτωση όλες τις επιχειρήσεις πέρα από ένα μέγεθος συγκεκριμένο, τότε θα βάλουμε κάποιες τιμές κατόφλια ούτω ώστε να μην καταλήξουμε να ζητάμε από κάθε επιχείρηση όλα αυτά τα καινούργια καθήκοντα, διότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε έναν κατακλυσμό ή σε ένα νεκροταφείο πληροφοριών και ε, στοιχείων που δεν θα, δεν θα χρησιμοποιούνται από κανέναν. Το θέμα είναι αν θα υποχρεώσουμε μια επιχείρηση τέτοια έργα να ε, αναφέρονται το κάθε ένα χωριστά και αναχώρα όπου δραστηριοποιείται και αν αυτό θα πρέπει να εξαρτηθεί από το μέγεθος της επιχείρησης, κύκλο εργασιών δηλαδή, από το μέγεθος του έργου και με βάση τις πληρωμές που γίνονται σε μια χώρα ή που βάσει ενός έργου πηγαίνουν προς την ε, κυβέρνηση ή την ε, τοπική αρχή. Αυτή την προσέγγιση εγώ την συζήτησα πολύ με τους σκιώδεις εισηγητές και διαπίστωσα από τις συζητήσεις μου ότι σε ορισμένα σημεία συμφωνούμε, αλλά σε πολλά σημεία που εγώ νομίζω σημαντικά, ακόμη δεν βρήκαμε μια συμφωνία. Να μπω σε κάποιες λεπτομέρειες. Είχα την εντύπωση συγκεκριμένα ότι με μια σειρά από εταιρείε θα πρέπει να αρχίσουμε π.χ. εξορυκτικές και επιχειρήσεις υλοτομίας. Να αρχίσουμε από αυτές είχα πει και πρότεινα πέραν τούτου ε, να συμπεριλάβουμε και μια κατηγορία μεγάλων αγροτών που τελευταία ε, είχαν ε, κατηγορηθεί ε, είχαν κατηγορηθεί α, και για, σκάνδαλα. Οι άλλοι συναδελφοί, με την εξαίρεση του ECR, θεωρούσαν ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε όλες τις επιχειρήσεις και από τη γαλακτοβιομηχανία και από την επεξεργασία τελειοποίησης κλπ. Θα μπορούσα να συμφωνήσω αν όντως θα εισαγάγαμε τιμές κατοφλίων που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα υποχρεώνεται κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθος ε, να δίνει αυτά τα στοιχεία. Και οι τιμές κατοφλίου ήταν οι εξή. Ότι πρέπει να έχουν τζίρο πάνω από 500 εκατομμύρια, τα έργα θα έπρεπε να ανέρχονται σε 25 εκατομμύρια ευρώ και οι πληρωμές προς τις κυβερνήσεις, είτε είναι φόροι, άλλες πληρωμές, παραχωρήσεις κλπ. θα πρέπει να ξεπερνούν τα, 100.000 ευρώ. Αυτές οι τιμές, οι οριακές που πρότεινα εγώ, θεωρήθηκαν σαφώς πολύ υψηλέ από τους συναδέλφους και οι αντιπροτάσεις τους ήταν, εις ό,τι αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων, κάθε επιχείρηση που είναι μεγαλύτερη από τον επίσημο ε, ε, ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης 1250 εργαζόμενοι 500 ε, τζίρο και όλες έπρεπε δηλαδή να υποβάλουν τέτοιες καταστάσεις. Για τα έργα είπαν οι συνάδελφοι όλα τα έργα. Λέω δεν είναι δυνατόν αν δηλαδή θα πρέπει να ασφαλτοστρωθεί ένα πάρκινγκ έργο είναι και αυτό και κάνει 6.000 ευρώ η κατασκευή του. Πρέπει να γίνει ε, κατάσταση και για αυτά και για τις πληρωμές προς τις κυβερνήσεις. Ε, είπαν 15 ή 20.000 και μόνο οι πράσινοι μίλησαν για 50.000. Εγώ είχα πει 100.000. Οπότε εδώ πόρο απέχουμε ακόμη από μια συμφωνία. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το ερώτημα αν οι πληροφορίες αυτές που θα δίνονται και εδώ πρόκειται για μία σειρά πληροφοριών, τζίρος, κόστος, συνεργάτες, φόροι κλπ, εργαζόμενοι δηλαδή φόροι κλπ, αν οι πληροφορίες αυτές θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ετήσιας ε, έκθεσης απολογισμού και αν θα πρέπει οι ορκωτοί ελεγκτές που θα εξετάζουν τους ισολογισμούς των εταιριών και τους ελέγχουν. Αν λοιπόν αυτά τα στοιχεία θα είναι κομμάτι του ετήσιου ισολογισμού που θα πρέπει επίσημα να εξετάζεται από τον ορκωτό λογιστή. Τώρα, αν συμβεί αυτό θα έχει τις εξής συνέπειες. Πρώτον, οι τέσσερις ε, μεγάλες ε, εταιρείες εργοτών λογιστών θα ε, τσιμενταριστούν, θα λέγαμε, ως ολιγοπόλια. Γιατί εκτός από τις τέσσερις μεγάλες, σε χώρες του τρίτου κόσμου δεν υπάρχουν άλλες. Αν αποφασίσει κάποιος να πάρει ορκωτό λογιστή, θα πρέπει να εξετάζει αυτός ο εργοτός λογιστής όλα τα έργα στις διάφορες χώρες. Άρα λοιπόν εδρεώνουμε την ολιγοπολιστική θέση των μεγάλων εταιριών ορκωτών λογιστών, πράγμα που δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχει και μια άλλη οδηγία που θέλουμε να πετύχουμε το άλλο πράγμα για τους οικονομικούς ελέγχους. Επίσης θα είναι πολύ μεγάλα τα παρεπόμενα ε, ε, ε, κόστη και μεγάλη γραφειοκρατική δαπάνη. Έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον για την αρχή και μετά από κάποιο διάστημα μπορεί να το αναθεωρήσουμε αυτό, να τα αλλάξουμε το... στην αρχή τουλάχιστον, να ε, συμβιβαστούμε με τα στοιχεία τα οποία ε, έτσι κι αλλιώς θα έχει μια επιχείρηση σε μια έκθεση διαχείρισης, γιατί μια χρηστή επιχείρηση έχει ε, σύστημα εσωτερικών ελέγχων που του δίνει τα βασικά στοιχεία αναχώρα και αναέργο που αναλαμβάνει. Και εδώ υπάρχει διαφορά. Όλοι οι άλλοι σκιώδεις θέλουν οι πληροφορίες αυτές επισήμως να αποτελούν κομμάτι του ετήσιου ισολογισμού των επιχειρήσεων και θα πρέπει να ε, καλύπτονται από τον έλεγχο του ορκωτού λογιστή. Αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η γνωμοδότησή μας είναι μόνο γνώμη η καθήλυν αρμόδια επιτροπή είναι η νομική επιτροπή, η οποία από ό,τι κατάλαβα ε, από συνομιλίες με τον ε, κύριο Λένε που είναι ο συγητής και το πρόεδρος της Επιτροπής ε, έχουν απόψεις εκεί πιο κοντινές με τις δικές μου από ότι με εκείνες των σκιωδών. Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε με τέτοια αυστηρότητα όπως ε, λένε οι σκιώδεις και που έχουν την πλειοψηφία δεν αμφισβητώ. Αν λοιπόν ακολουθήσουμε την αυστηρότητα των σκιωδών, διατρέχουμε τον κίνδυνο η γνωμοδότησή μας να μην ληφθεί υπόψη από την Νομική Επιτροπή. Και για να τελειώσω, ε, μερικές παρατηρήσεις ακόμα. Η Πράσινη και ο συνάδελφος Φέρμπερ από το ΕΛΚ πρότειναν να διαγράψουμε τα άρθρα 6 και 7 που πρόκειται για το fair value, ε, την δίκαιη αξία. Εγώ νομίζω ότι η αξιολόγηση των χρηματοδοτικών μέσων θα πρέπει να στηρίζονται στο fair value, όπως και παλιότερα, διότι αλλιώς ε, τα ε, χρηματοπιστωτικά μέσα που κυμαίνονται πολύ στην αξία τους, έχουν μεγάλη διακύμανση και που κάποια στιγμή συρρυκνώνονται σε σχέση με την τιμή κτίσεως, ε, αξιολογούνται λάθος και η τιμή που θα παρουσιάζεται θα είναι ε, λάθος, θα είναι ψεύτικη. Το είδαμε και στα κρατικά ομόλογα. Επίσης, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην επίσημη, πρέπει να μείνουμε στην επίσημη ταξινόμηση της Κομισιόν και όχι να πούμε, όπως λέει ο κύριος Μίτσελ, ε, να έχουμε δύο, δηλαδή τζίρο και ισολογισμό. Τέλος, έχω ε, προσθέσει κάτι που δεν υπήρχε στην πρόταση της Κομισιόν, ότι δηλαδή ε, τις εισηγμένες εταιρείες, α, τις εισηγμένες και όλες τις ε, που λειτουργούν με βάση και ε, υποβάλλουν ισολογισμό με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, αυτές οι δύο κατηγορίες επιχειρήσεων στο μέλλον θα υποχρεώνονται να, ε, βάλ, να εισάγουν ε, ηλεκτρονική ε, ε, έκθεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Διότι έτσι θα έχουμε μια κοινή βάση για να συλλέγονται οι πληροφορίες από όλε τις επιχειρήσεις με τρόπο γρήγορο. Και θα είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι συμβατές οι πληροφορίες. Ε, δηλαδή οι εφορίες, ε, κτηματολόγια, στατιστικές υπηρεσίες να έχουν έναν ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστώ τον Βολφ Κλίντ ε, και του Σκιώδη. Η μέθοδο εργασία μου οδηγεί συνήθω σε συνένεση. Κάτι το οποίο είμαστε αρκετά δυνατοί εδώ στο Κοινοβούλιο. Τώρα. Πολλά από τα ζητήματα που έθεσε ο συνάδελφος Κλίντ ε, παραμένουν ακόμα ανοιχτά. Προτού να εξετάσουμε αναχώρα, να πω ότι είναι πολύ επίμαχο το ζήτημα. Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα πολύ σημαντικά ε, αφορούν στην οδηγία διαφάνειας. Ε, τώρα, όταν πρόκειται για ορισμούς, οι προτάσεις ε, νομίζω πως είναι κατάλληλες. Ε, η Κομισιόν θα πρέπει να υποβάλει μια έκθεση στο μέλλον η οποία θα αναλύει τις ε, διάφορες επιλογές αναφορικά με τους ορισμούς τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι σημαντικό. Θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση σε ό,τι φορά την έννοια αυτών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ένα ζήτημα το οποίο παραμένει ανοιχτό. Υπάρχουν αντιφατικές τροπολογίες για τις εκθέσεις οι οποίες θα πρέπει να δημοσιεύονται. Υπάρχει πρόταση ότι αυτό θα αναφέρει φορά μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. και αυτό φυσικά θα πρέπει να το αποφασίσουν τα κρατη αλλά θα πρέπει και εμείς να το εξετάσουμε περαιτέρω και να το σχολιάσουμε. Τώρα ένα δεύτερο ζήτημα είναι η εναρμόνιση τα κράτη-μέλη μπορούν να έχουν απαιτήσει πιο αυστηρές από αυτέ που περιέχονται στην οδηγία. Υπάρχουν και εδώ κάποιες αντιφατικέ προτάσει. πρόθεσή μου είναι να συμφωνήσω με την πρόεδρο τη Κομισιόν σχετικά με τις απαιτήσει υποβολής εκθέσεων. Ένα άλλο ζήτημα είναι η εναρμονισμένη ηλεκτρονική αναφορά εκθέσεων και το Accessible Business Reporting. Εγώ θα ήμουν υπέρ μεν, αλλά ας δούμε αν μπορέσουμε να βρούμε κάποιου συμβασμού στο πλαίσιο των πολιτικών μας ομάδων. Και κάτι ακόμα και θα ήθελα εδώ σχολιασμό από τους συναδέλφους σου. και αναφέρομαι στους τρόπους ε, υπολογισμού των ε, δικαιωμάτων ψήφου. Φυσικά αυτό αφορά ε, τους ψήφους των μετόχων τώρα. Όπως είπε ο Κλίντ, ο Κλίντ έχει Υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα εκτός από την ECR και την ALDE. Και μιλάμε για τους ορισμούς, για το πεδίο εφαρμογής, για το ποιες τα αναφέρουν και όχι μόνο οι εξορυκτικές και οι επιχειρήσεις υλοτομίας, να συμπεριφθούν και άλλοι κλάδοι. Και ξέρουμε ότι οι οι εταιρείε οι οποίε δεν είναι εισαγωγμένε στην στη διαπραγμάτευση μπορούν να οδηγήσουν σε ε, προβλήματα στον τομέα του ανταγωνισμού, δηλαδή σε του ανταγωνισμού μπορούμε νομίζω να μπορούμε να βρούμε κάποια συμβασμούς εδώ. Τώρα, ά δύο θέματα. Το ένα θα έπρεπε να αποτελούν ε, θέμα των ε, ελέγχων. Τώρα επίσης το ζήτημα των ε, θέσης των Γερμανών για τα κατόφλια και υπάρχει και μια άποψη με την οποία συμφωνούν συμφωνεί ένα σημαντικό κομμάτι των πολιτικών κομμάτων θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο έλεγχος των οικονομικών δεν ξέρουμε πόσο άχθος θα προκαλέσει ένας τέτοιος έλεγχος για τις επιχειρήσεις αλλά μεγάλες ε, ελεγκτικές εταιρείες ελέγχουν τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε ότι δημιουργούνται κάποιες ε, μονοπωλιακές, ε, ολιγοπωλιακές καταστάσεις με τις οποίες κανείς δεν συμφωνεί. Έχουμε ακούσει σχόλια και επιχειρήματα υπέρ και κατά. Αλλά το βασικό επιχείρημα είναι ότι αν αυτό ο έλεγχος εμπίπτει στο πλαίσιο του υποβολής αναφορών, μιλάμε για ένα soft reporting και υπάρχουν φυσικά νομικές ε, επιπτώσεις εάν αυτές οι εκθέσεις ε, δεν είναι ορθές. Ε, εντάξει, πάντα μπορεί να πει κάποιο ότι παρερμήνευσα κάποια στοιχεία, έγινε λάθος κλπ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για διαφάνεια, την οποία θέλουμε να πετύχουμε. και έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα ελέγχων και υπάρχει μια δεσμευτική δομή διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν ε, ε, επιβάλλουμε κυρώσεις στην επιχείρηση για τις συναλλαγές αλλά μόνο για θέματα αστικής ευθύνης. Και ο έλεγχος θα πρέπει να διεξάγεται. Διαφορετικά χάνει κάθε νόημα η όλη προσπάθεια που καταβάλουμε. Τώρα τα κατόφλια. Υπάρχουν τριών ειδών. Το μέγεθος των επιχειρήσεων, που θα πρέπει να βάλουν εκθέσεις, νομίζω ότι υπάρχει ευρύτατη συνένεση ότι το όριο θα πρέπει να είναι το όριο των κομισιών επιχειρήσεων. υπάρχουν διστάμενες απόψεις σχετικά αν θα πρέπει να είναι το επίπεδο, το των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή το διπλάσιο ή το τριπλάσιο ή το δεκαπλάσιο που ήταν η αρχική θέση του κυρίου Κλίντ. θέση μου, όπως και θέση των υπολείπων ομάδων πριν της άλτε ήταν να παραμείνουμε τον ορισμό των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το διπλάσιο-τριπλάσιο, δηλαδή 100 εκατομμύρια. Αλλά δεν έχουμε ακόμα πετύχει συμφωνία. Τώρα για τα κατόπια των πληρωμών, ε, εδώ έχουμε μεγαλύτερη, μικρότερη μάλλον ευελιξία, διότι αν λάβετε τα 2.000 ευρώ από πλευρά επιχείρηση είναι ένα χαμηλό ποσό. Αλλά εάν το δείτε από πλευρά της ε, χώρας, της ανεψόμενης χώρας των μισθών των υπαλλήλων 20.000 ε, ευρώ είναι πολλά χρήματα και μπορεί να έχουν επιπτώσει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα ήθελα να διατηρηθεί το κατόφλι ε, ή δυνατόν χαμηλότερα. Και το τρίτο σημείο είναι η υποβολή εκθέσεων κάθε άδεια και κάθε, κάθε, κάθε σύμβαση θα πρέπει να αναφέρεται για συμπεριλαμβάνεται στις ετήσιες εκθέσεις αλλά εδώ θα πρέπει να έχουμε κάποιο χαμηλό όριο 10.000 ευρώ και μια νέα διατύπωση η οποία περιγράφει ότι δεν θέλουμε να αποφύγουμε να μην έχουμε ψηλά κατόφυλλα όπως η δασική βιομηχανία που έχουμε 500.000 ευρώ έργα για υλοτόμηση δασών και θέλουμε να αποφύγουμε να γίνεται ε, κατα, κατάτμιση των δασών σε μικρά κομμάτια για να αποφεύγονται οι υποχρεώσεις που επιβάλλει η νομοθεσία και κάτι ακόμα ειδικά με το Συμβούλιο και τις διαπραγματεύσεις, ε, γνωρίζοντας πώς έχει κατάσταση το Συμβούλιο, θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα σαφείς ε, πάνω στο ζήτημα αυτό, διότι ούτως ή άλλως θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις και πρέπει να υπάρχει χώρος ε, για να υπαναχωρήσουν ενδεχομένω. Ευχαριστώ. Αυτή, αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλο από ό,τι βλέπουμε. Υπάρχουν δέκα σκιώδεις, Δέκα σκιώδεις, μεγάλη γνωμοδότηση. Πρώτα, ο Μισελ Γκέι. Δεν είναι εδώ, κύριος Μπούλμεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα μιλήσω για λογαριασμό του συναδέλφου Έντβαρτ Σικλούνα. Γιατί δυστυχώς δεν μπορούσε να έρθει. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην επίλυση του προβλήματος εμείς οι σοσιαλδημοκράτες. Έχουμε παρόμοια θέση και στις δύο εκθέσεις. Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές και τον Βολφ Κλίντς και την Τσέρβα Πιετικάινεν για την εξαιρετική δουλειά που μας δίνει μια βάση για τις συμβιβαστικές διαπραγματεύσεις που τώρα θα τελειώσουν. Καταρχήν μια πολιτικής φύσεως παρατήρηση για να μην χαθούμε στις λεπτομέρειες και στις αποχρώσεις ε, του θέματος. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε. Εμείς όταν είμαστε εταίροι άλλων χωρών, ιδιαίτερα χωρών του Νότου, των χωρών ΑΚΕ κλπ. Συνήθως μιλάμε για καλή διακυβέρνηση, good governance. Θέλουμε από τα κράτη εταίρους μας ακέραιη συμπεριφορά, διαφάνεια στη συμπεριφορά, ε, σύγχρονες κρατικές μορφές. Εκεί όπου έχουμε αποκτήσει περισσότερες εξουσίες από τη συνθήκη της Λισαβόνας και τώρα στο εξωτερικό εμπόριο μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα στα πλαίσια της συναπόφασης. Προσπαθούμε να καταρτίζουμε συμβάσεις δίκαιες, ε, σωστές, όπου ε, σημαντικά θα είναι τα ποιοτικά κριτήρια και όχι η εσπευσμένη δράση. Τώρα, με τις δύο εκθέσεις των δύο συναδέλφων, θέλουμε να μιλήσουμε για οικονομικές καταστάσεις που πρέπει να υποβάλλονται, διαφάνεια στην επιχειρηματική συμπεριφορά και θα πρέπει να λειτουργήσουμε με τα ίδια κριτήρια και τις ε, αρχές. Θέλουμε καθαρές συναλλαγές θέλουμε ε, να διατηρήσουμε τον θεμητό ανταγωνισμό. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, κλίμα εμπιστοσύνη στη διεθνή οικονομική κοινότητα. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε με λόγια καθαρά στους δύο, στις δύο εκθέσεις, να μην συμβιβαστούμε με τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, αλλά να προχωρήσουμε με στόχους φιλόδοξους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην προσέγγιση country by country, αναχώρα, που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις και θα πρέπει να δούμε πολύ συγκεκριμένα τις πληρωμές, να μην είμαστε υπερβολικά γενναιόδοροι με τις εξαιρέσεις μας και να προσανατολιστούμε προς τον ορισμό των ΜΜΕ όπως ήθιστε στα άλλα νομοθετήματα. Δεν νομίζω ότι πρέπει εδώ να αποδυναμώσουμε το κείμενο. Ε, δεν συμφωνώ ε, να υποχωρήσουμε εδώ. Καταρχήν θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια επιχειρηματική κουλτούρα η οποία δεν θα επιβαρύνει τις ΜΜΕ αλλά που θα υποχρεώνει τις μεγάλες τις προδιαγραφές που θα αποφασίσουμε. Δεν θέλουμε ειδική έκθεση, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει νομίζω ότι θα πρέπει να μπαίνει στον ετήσιο ισολογισμό. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό γιατί μπορούν έτσι αν χρειαστεί να υπάρξουν και νομικές επιπτώσεις αν διαπιστωθεί κάποια ε, απάτη ή πρόβλημα. Ε, βλέπω ότι οι περισσότεροι σκιώδεις είναι υπέρ της φιλόδοξης προσέγγισης και νομίζω ότι ε, και η Επιτροπή ΕΚΟΝ θα συμφωνούσε με μια τέτοια προσέγγιση και έτσι ενδεχομένως και οι πιο διστακτικοί ανάμεσά μας κάποια στιγμή θα πιστούν ότι είναι σωστό να προχωρήσουμε με πιο φιλόδοξο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Uh, uh, θα είμαι πολύ σύντομο Ρωτήσα καν και ούντο, οι προλαλήσαντε είπαν αυτά τα οποία, με τα οποία συμφωνούμε, γιατί αυτό είναι περιττό να επαναλάβω τα ίδια. Αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό και καταλαβαίνω ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε πολύ μεγάλο βάρος στις επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να αναζητήσουμε ποιο θα είναι το όφελο σε σχέση με το κόστος. Δεν είναι απλά και μόνο κάτι το οποίο οδηγεί σε επιπλέον δαπάνες αλλά και σε επιπλέον ωφέλη. Αν κάνω μια αναδρομή στο παρελθόν, στα 15 προηγούμενα χρόνια, ορισμένε ε, επιχειρήσεις είχαν άλλες διαδικασίες ε, για να βρουν νέε εργασίες στην αγορά. Τώρα είναι πολύ πιο δύσκολο να υπάρξει κάτι το καινούριο στην αγορά. Αλλά ένα καινούριο φάρμακο, α πούμε, αλλά υπάρχει ασφάλεια των φαρμάκων. Έτσι μπορεί κανεί να δικαιολογήσει την επιπλέον δαπάνη του εγχειρήματο το οποίο σημαίνει περισσότερη δουλειά. Και αν θέλουμε αυτά τα στοιχεία να είναι ε, σωστά και αξιόπιστα, σημαίνει περισσότερη δουλειά και περισσότερη δουλειά και για του ελεγκτές. Αν θέλετε λοιπόν μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη, έτσι υπάρχει ανάπτυξη. Αν θέλετε περισσότερε δουλειέ, έτσι θα βρεθούν περισσότερε δουλειέ. Αστείευομαι. Όσον αφορά όμω ε, το κατόφλι των επιχειρήσεων, ό,τι κάναμε το CCCTB ε, θα μπορούσα να πω εντάξει ω ένα πρώτο βήμα συμφωνούμε για το διπλό επίπεδο σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μετά αν η πρώτη φάση ε, στεφθεί με επιτυχία θα περάσουμε στη δεύτερη φάση. Καταρχήν όμως αυτή, ε, αυτός θα πρέπει να είναι ο κανονικός τρόπος ε, που θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Δεν θα πω περισσότερα για τα κατόφλια και ζητώ συγγνώμη που είμαι τόσο βιαστικός, αλλά έχω ανηλυμένες υποχρεώσεις άλλες. Ευχαριστώ. Ε, yes, Mr. President, I... Πρόεδρε, και εγώ θα μιλήσω εξ ονόματος ε, Majesty the Queen's Jubilee το Φταμάλ που βρίσκεται ε, στο Ιωβιλέο της Βασίλισσας. Όχι, εδώ είναι ακόμη, δεν, είναι, δεν έχει φύγει. Okay. I'll tell him. I'm going check him out. Mr. Um, President... Κύριε Πρόεδρε, όταν συζητήθηκε αυτή η γνωμοδότηση τελευταία φορά, συμφώνησα να γίνει μια αναθεώρηση των οδηγιών, ε, οι οποίες υπάρχουν εδώ και 30 χρόνια, να περιοριστεί η γραφειοκρατία, να υπάρχει μεγαλύτερη συγκρισιμότητα ε, και να υπάρχει ένα τίμιο παιχνίδι, ώστε οι επιχειρήσεις να βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιριών. Τώρα, όσον αφορά την, ε, την αναφορά των πληρωμών στις κυβερνήσει, πρέπει να βρεθεί μια σωστή ισορροπία μεταξύ των αναγκών διαφάνεια και του υπερβολικού βάρου για τι επιχειρήσει. Σήμερα θα αναφερθώ σε δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα την αναφορά χώρα προς χώρα. Αναχώρα. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ με την αρχή αυτή τη αναφορά αναχώρα για τι εξορρυκτικέ βιομηχανίε. Το γεγονό ότι τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή επίση συμφωνούν είναι μια κατάσταση που χαιρετίζουμε. Αλλά απογοητεύουμε από το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο μάλλον σπρώχνει πολύ και με ριζικό τρόπο για να προσαρμόσει αυτή την αρχική πρόταση χωρίς να έχουν γίνει εκτιμήσεις επιπτώσεων. Και αφήνει περιθώριο σε όλες τις επιχειρήσεις ε, προσπαθώντας να καθορίσει τι είναι το project, τι κάνει, τελικά επιβραδύνει τη διαδικασία. Και φοβούμαι ότι αυτό το οποίο θα μπορούσε να ε, συμφωνηθεί μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες θα απαιτηθούν τώρα πολλά χρόνια. Δεύτερον, όσον αφορά τις ε, τροπολογίες που κατέθεσα εγώ και ο κ. Καμάλ για την τίμια και δίκαιη αρχή, πιστεύω ότι είναι ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα και στην Επιτροπή και ε, στο Συμβούλιο ε, Διεθνών Προδιαγραφών. Διότι θα πρέπει να βασίζονται οι κανόνες όχι μόνο στη σύνεση αλλά και στην πραγματικότητα παρά το γεγονός ότι αυτή η οδηγία δεν αφορά μόνο την εφαρμογή του FAS μπορούμε όμως με αυτή την ευκαιρία να διευκρινίσουμε ε, τι σημαίνει η δίκαια αρχή. Η Επιτροπή ε, λάθος ε, συμπεραίνει ότι αυτή η αρχή ε, ε, αυτή η αρχή είναι μια ουσιαστική αρχή, η οποία, το οποίο κατέστησε σαφέ από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 1996 και το 99. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ορισμένε προδιαγραφές κανόνες ε, αναφοράς δεν επιτρέπουν στις τράπεζες να παρουσιάσουν τους λογαριασμούς με τρόπο που θα είχε αποφευχθεί και αυτό προς το συμφέρον μας. sorry. Uh, I'm trying to see προσπαθώ να δω αν και άλλοι σκιώδεις είναι εδώ. Ο κύριος Σέπινγκ μίλησε, εκπροσωπήθηκε. Μιλήσατε και για λογαριασμό του κυρίου Καμάλ και του κυρίου Έπινγκ. Ο κύριος Χάγκλουντ δεν είναι εδώ. Και ο κύριος Κλούτε δεν είναι εδώ. Καλώς. Δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Μακάρτιν. Δεν έχω την ίδια κρυστάλλινη μπάλα ε, όπως έχει ο συνάδελφος. Ε, θα μπορούσαμε ίσως να είχα, πρέπει να περιμένουμε ίσως αρκετά χρόνια όπως λέει. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό το θέμα τελικά είναι τόσο σημαντικό για μας και οι λεπτομέρειες είναι σημαντικές και αυτή η αναφορά αναχώρα είναι επίσης σημαντική και τελικά θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι αντικατοπτρίζουμε και τις απόψεις αυτής της Επιτροπής και όπως δείχνουν οι συζητήσεις και τις 165 τροπολογίες που καταθέτηκαν, ε, κατατέθησαν στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Γι' αυτό, ως ο δημοκρατικός θεσμός, θα πρέπει να δεχθούμε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους ε, ψηφοφόρους μας και τις οργανώσεις εκτός του Κοινοβουλίου και δεν μπορούμε να το δούμε πρόχειρα λέγοντας ότι απλά και μόνο δεχόμαστε ε, τις θέσεις τις οποίες έχει εκφράσει η Προεδρία της Δανίας. Παρόλο που μπορεί να είναι καλές αυτές οι θέσεις, πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να τηρούμε τις δημοκρατικές αρχές, διότι αυτή η οδηγία αφορά τη διαφάνεια. Λοιπόν, εμείς πρέπει να επιδεικνύουμε διαφάνεια όσον αφορά την αντιμετώπιση των θεμάτων μας. Με τα χαράς, λοιπόν, θα δεχθώ ε, τις προτάσεις της Επιτροπής ΕΚΟΝ, διότι νομίζω ότι είναι σημαντική συμβολή στο έργο ε, των εισηγητών και απλά θα ήθελα να κάνω μερικές ε, μικρές παρατηρήσεις, ε, διότι πρέπει να δούμε τι θα συμφωνηθεί μεταξύ των σιωδών. Είναι σαφές, ε, όταν βλέπω τις τροπολογίες, ότι θα πρέπει να περιληφθούν στην ετήσια έκθεση, διότι εκεί, από εκεί προέρχονται οι περισσότερες τροπολογίες. Και αν θέλουμε να έχουμε μια σωστή προσέγγιση, ελέγχθη ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. Γι' αυτό θα ήταν λάθος για μας να ακολουθήσουμε άλλη μέθοδο, κυρίως εάν δεν υπάρχει εναλλακτική προσέγγιση η οποία να, είναι, να λειτουργεί, να είναι σωστή. Δεν βλέπω άλλες επιλογές, σε πάση περιπτώσει. Επίσης πιστεύω ότι όλο αυτό το θέμα για το κόστος και τα λοιπά είναι σημαντικό να το δούμε, να το σκεφτούμε. Αλλά ο Λόρντ Μπράιν, πρώην ε, πρόεδρος της BP, έλεγε ότι δεν είναι τόσο δύσκολο για τις μεγάλες εταιρείε να το κάνουν, διότι ήδη συλλέγουν τις πληροφορίες αυτές και το επιπλέον κόστος θα ήταν αμεληταίο. Λοιπόν, αυτό το είπε κάποιος ο οποίος βρίσκεται στον κλάδο. Και μιλάμε για τις εξωτερικέ βιομηχανίες και την αναφορά χώρα προς χώρα. Ναι, το ξέρω. Πρέπει όμω να διαπραγματευτούμε ορισμένα θέματα. Γι' αυτό οι μεγάλε εταιρείε, οι μεγάλε επιχειρήσει μπορούν να το κάνουν. Ναι, αυτό είναι φανερό σε κάθε κλάδο. Και δεν έγινε μια τελική συζήτηση για το τι θα κάνουμε με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αυτό πρέπει να συζητηθεί ακόμα. Νομίζω λοιπόν ότι σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση να γίνει τέτοια αναφορά ενώ το Συμβούλιο δεν το λέει αυτό. Λέει το επίπεδο της κυβερνητικής αναφοράς. Και επίσης αυτό είναι ουσιαστικό σε χώρες όπως, στην Αφρική για παράδειγμα, τα εισοδήματα είναι έξι φορές μεγαλύτερα από τις εξορρυκτικές βιομηχανίες από ότι είναι ε, ε, το εισόδημα που προέρχεται από τη βοήθεια στην ανάπτυξη στην Ουγγάντα έχουν δισεκατομμύρια από τις εξορρεκτικές βιομηχανίες. Μιλάμε λοιπόν για πολλά χρήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, σαφήνεια, ώστε αυτές οι χώρες να καταπολεμήσουν τη διαφθορά, να γνωρίζουν πού πηγαίνουν τα χρήματα και νομίζω ότι μας παρουσιάζεται, μας δίνεται μια ευκαιρία σε αυτή την έκθεση. Δεν μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και να το ξαναδούμε αργότερα να αναθεωρήσουμε τη θέση μας ε, για να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Συνεπώς θα πρέπει να είμαστε πιο ριζικοί, ε, να διαπραγματευτούμε πολύ με την Επιτροπή, να δούμε τι θα επιτύχουμε. Τώρα, πιο τεχνικά θέματα, όπως είπα, και άλλα πρέπει να γίνουν από την Επιτροπή μας ε, και αναμένω το αποτέλεσμα. Είχα όμως μια συζήτηση με τον κύριο Κλίντς σχετικά με το XPRL, το θέμα κατά πόσον αυτό, αυτή, αυτό, αυτή η προδιαγραφή, αυτό ο κανόνας πρέπει να είναι υποχρεωτικός. Και γνωρίζω ότι και η Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων ζητάει αυτό ο κανόνα είναι υποχρεωτικό. Δεν ξέρω αν πρέπει να επιβάλλουμε προδιαγραφέ πρότυπα σε αυτό το τομέα. Ε, δεν, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πρότυπα και κανόνε βιομηχανίε. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Ε, ας πούμε εφαρμόζουν ε, με βάση το XPRLL και το XBRL που μπορεί να έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Νομίζω ότι αν δούμε τις έρευνες που έχουν γίνει, ε, δεν καταλήγουν πουθενά, δηλαδή δεν καταλήγουν στο ότι η XBRL είναι η καλύτερη προσέγγιση. Το άλλο θέμα είναι ότι και ΣΜΑΡ επίση το εξετάζει, κοιτάει την ανάλυση κόστους ωφέλους για να δει κατά πόσον αυτή είναι η καλύτερη λύση. Ακόμα και στις ΗΠΑ δεν έχει επιβληθεί, αλλά είναι εθελοντική αυτή η λύση. Δηλαδή μπορούν να κάνουν αναφορές εταιρείε με βάση το XBRL. Μπορούν να το κάνουν εθελοντικά χωρίς να είναι υποχρεωτικό. Λοιπόν, μπορούμε και εμείς να, να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση, ανάλογα με την, την έκβαση της ψηφοφορίας σα. Δεν πρέπει να σπρώχνουμε προ την υιοθέτηση του XBRL μπορούν, αν θέλουν, ε, προαιρετικά να υιοθετήσουν αυτή τη μέθοδο και αν χρησιμοποιηθεί περισσότερο αυτή η μέθοδος, τελικά θα γίνει το πρότυπο, ε, ε, ο κανόνας που θα χρησιμοποιεί η βιομηχανία. Αν είναι ευρέως διαδεδομένο. Αλλά αναμένουμε με υπομονησία τις προτάσεις σας ε, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Δεν το συζητήσαμε εδώ, γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Η Επιτροπή χρησιμοποίησε την, άκτα και νομίζω ότι αυτό είναι λυπηρό, επειδή δεν είχαμε ακόμα μια επίσημη συζήτηση, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια γνωμοδότηση από την Επιτροπή και να μην γίνονται συνέχεια συζητήσεις. Άτυπα θα συζητήσουμε με την Προεδρία αυτά τα θέματα, αλλά όπως είπα δεν είμαστε εξουσιοδοτημένοι. Γιατί πρέπει να συζητήσουμε πρώτα τι ε, τροπολογίε που έχουν κατατεθεί. Και ε, τελειώνει αυτή η Προεδρία, δεν θα έχουμε χρόνο μετά υπάρχουν οι καλοκαιρινέ διακοπέ, δεν θα υπάρχει χρόνο. Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα μέσα στι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Αλλά αναμένω ε, τη γνωμοδότηση από την Επιτροπή σα Ευχαριστώ. If uh, nobody else is... Αν ε, δεν επιθυμεί κάποιο άλλο συνάδελφο να λάβει το λόγο, δώσω το λόγο στον κύριο Κλίντ και στην κυρία Πίτερ Κάινα. Δεν έχω πολλά να πω. Ευχαριστώ τους Κιώδης ε, και την Αρλίν για την συμβολή της. Ε. Σε κάποιους τομείς διαφωνούμε. Θα δούμε μέσα στις επόμενες μέρες ε, αν μπορούμε να γεφυρώσουμε το κενό. και θα ήθελα να το συζητήσω το ζήτημα στην πολιτική μου ομάδα την επόμενη εβδομάδα και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να συγκλίνουμε και να καλύψουμε το χάσμα. Δεν χρειάζεται σε αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή να έχουμε μια κοινή άποψη, αλλά απλά πρέπει να έχουμε μια θέση για να μπορούμε να μεταβούμε στον τριμερή διάλογο μια θέση η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα, μια θέση προς ε, συζήτηση με το Συμβούλιο να μην μας πει μα εσείς αυτά που λέτε είναι παρανοϊκά δεν μπορούμε να καθίσουμε για τραπέζι και να τα συζητήσουμε δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο αλλά εμείς τόσοι εκφύσεως είμαι αισιόδοξο δεν απογοητεύομαι κυρία Πίτη είναι α, ο κύριος Κλίντς το XBRL θα θέλαμε να το περιορίσουμε στις ε, επιχειρήσεις που εφαρμόζουν IBRS. Δεν ε, έχουμε επίση και ένα χρονοδιάγραμμα κατά νου που αφορά στο 2018. Τώρα, σχετικά με τις... Ε, θα ήθελα να ακούσω την Κομισιόν πριν από την τελευταία μου παρέμβαση. Δεν ξέρω αν ο πρόσωπος της Κομισιόν θέλει να πει κάτι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα τα οποία τέθησαν. Δεν θα ήθελα να μπω σε μια γενική ζήτηση, αλλά να πω, όπως και ο κύριος Μπούμαν είπε, θα πρέπει να δούμε το συνολικό στόχο της πρότασης της Κομισιόν και ο στόχος ήταν να δημιουργήσει διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις στον εξωτερικό τομέα και στον, σε άλλους ε, μεγάλους κλάδους, σημαντικούς κλάδους. Ε, φυσικά θέλουμε να εξετάσουμε πώς μπορεί να πετυχθεί η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Θέλουμε να υπάρχει πραγματική διαφάνεια. Πρόκειται και για ένα ζήτημα ισορροπίων ε, σε ό,τι την τις επιχειρήσεις. Αν έχετε κατά νου μια επιχείρηση όπως η Shell, αυτή καταβάλει ένα δις ε, δολάρια ε, τα οποία είναι τεράστια ποσά ε, για σας για μένα και τι όμως διαφάνεια επιτυχάνεται ίσως όχι και πολύ τώρα συγκεκριμένο ερώτημα με τέθη σχετικά με τις ελέγχους αυτών των εκθέσεων να επιστήσω την προσοχή ότι ούτε στο σύστημα EITI που αναπτύχθηκε τα τελευταία 10 χρόνια, ούτε στο US.frank υπάρχουν σχετικές, ε, σχετικές απαιτήσει. Γιατί, διότι όλα αυτά τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν ε, ελέγχθηκαν μέσω των, του ελέγχου των λογαριασμών. Αν χρησιμοποιήσετε λοιπόν περαιτέρω απαιτήσει για αυτού του είδους τις εκθέσεις, τότε θα διπλασιάσουμε την εργασία και θα αυξήσουμε το κόστος. Η Κομισιόν φυσικά προσπάθησε να δημιουργήσει ένα ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού. Δεν θέλω να πούμε σε λεπτομέρειες, αλλά δεν θα θέλαμε να ακολουθήσουμε εντελώς διαφορετικό δρόμο από αυτόν που ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι μια προσπάθεια ε, απλούστευσης. Ε, έχουμε πετύχει μεγάλη πρόοδο απλουστεύοντας τους κανόνες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό θα είναι ένα από τα καλά στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις να έχουν ε, μικρότερο άχθος σε so XBRL πιστεύω φυσικά θα πρέπει να το ελέγξω αλλά έχουμε μια θετική άποψη περί αυτού. Έχει νόημα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τον IVRS και να το πράττουν και ηλεκτρονικά. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε μόνο επί χάρτου, αλλά όπως είπε και ο εισηγητής, έχει νόημα να γίνει ένας ε, διπλός έλεγχος ε, και είμαστε λοιπόν πολύ ανοιχτοί σε αυτό και το ποια θα είναι τελική μορφή βρίσκεται στα χέρια του Κοινοβουλίου και τέλος τώρα στην ε, ειλικρίνεια κοιτάξτε αυτό υπάρχει ήδη εδώ και 30 χρόνια είναι μια αρχή δώσαμε μεγαλύτερη έμφαση για αυτήν την ε, ειλικρίνεια, τη σαφήνεια. Οι λογαριασμοί θα πρέπει να είναι ανοιχτοί, καθαροί, σαφείς, να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τι βρίσκεται πίσω από τα στοιχεία, από τους λογαριασμούς τους. Και θέλουμε να δώσουμε ε, μεγάλη σημασία στην την έννοια της, ε, του ελέγχου και να είμαστε βέβαιοι ότι οι έλεγχοι αυτοί γίνονται με τον σωστό τρόπο και τα στοιχεία μιλάνε την αλήθεια. Τώρα σε, ό,τι αφορά τους ψήφους, απάντηση εκτός μικροφώνου. Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση για τη συνάδελφος ε, είναι η για αυτά τα δικαιώματα ψήφου. Το θέμα είναι ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό ε, των δικαιωμάτων ψήφου, η ονομαστική ή η δέλτα η πρόταση ήταν να επεκταθεί η Δέλτα σε όλα και μια άλλη